Otwieram posiedzenie. Podczas głosowania na wczorajszym posiedzeniu i artykułu 50 regulaminu Parlamentu Europejskiego przyjęto przez Συνεδρίαση βάσει του άρθρου 56 και 57 του κανονισμού. Αναφέρθηκε, ζητήθηκε, μάλλον έγινε επίκληση του άρθρου 56-57 του κανονισμού. είδαμε ότι δεν έγινε καμία προσφυγή βάσει του άρθρου 211 παράγραφος 4 του κανονισμού, άρα η ερμηνεία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στην συνάντησή της 14 Φεβρουαρίου του 2001 εγκρίνεται. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, των άρθρων 56 και 57, φεύγει από την ημερήσια διάταξη η έκθεση Ματιέ. Πρόκειται για ένα θέμα που συζητήθηκε επί μακρόν, τώρα υπάρχει μια σαφέστατη νομική εξήγηση. Η μερίσια διάταξη τώρα, α πούμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε καταρχά την δήλωση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την έκθεση προόδου 2010 σχετικά με την Κροατία. Συναντηθήκαμε χτες με τον Κροάτη Πρωθυπουργό, παρουσία και του κυρίου Σβόμποντα, και του Προέδρου της, ε, της αντιπροσωπείας με την Κροατία. Συζητήσαμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων της Κροατίας με την Ένωση και με μεγάλη ικανοποίηση σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να ε, παρουσιάσουμε το μέλλον της χώρας αυτής στο πλαίσιο αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία εδώ του Επιτρόπου κ. Φούλε και ζητώ από τον Προεδρεύοντα κ. Μαρτώνη να λάβει το λόγο εξ του Συμβουλίου. Γνωρίζουμε τη σημασία που δίδει η Ουγγαρία στο ζήτημα της ένταξης και σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο, κύριε Προεδρεόντα. Κύριε Μάρτονη. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εξ ονόματο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνομαι στην Ολομέλεια με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά σήμερα. Η συνάντηση